Σώτιμες κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι μια ιδιαίτερη τιμή για μένα να δώσω στην ε, κυρία Λαμία Χατζή Μπασάρ και την ε, Νάντια Μουράτ να τους πω το καλώς δύο πραγματικά εξαίρετες, ε, ξεχωριστές νεαρές ε, γυναίκες από ε, την κοινότητα των Ιωσίτα, οι οποίες, στις οποίες σήμερα απονέμεται το βραβείο Ζαχάροφ. Καλώς ορίσατε. Παρακαλώ Αγαπητοί συνάδελφοι, να καθίσετε στις θέσεις σας και καταρχήν εισαγωγικά να δείτε ένα σύντομο, μια σύντομη βιντεοτενία.